Τώρα έχουμε... ο κύριος Άλβες ζητάει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι. Η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού αξιολόγησε τα διαπιστευτήρια της κυρίας Μπετίνα Μισελ Ιάκοψεν, υποψηφίου για συμμετοχή στο ελεκτικό συνέδριο που είχε προβάλει το Συμβούλιο. Στη συνεδρίαση της 7ης Ιουνίου. Η κυρία Ιάκοψιν έχει σταδιοδρομία και επαγγελματικό υπόβαθρο ικανοποιητικό. Από το 2005 ήταν και εισηγήτρια στο Ελεκτικό Συνέδριο της Δανίας. Έχει επαγγελματική ανεξαρτησία και ακαιρεότητα ουδετερότητα. Οι ικανότητες αυτές λοιπόν και τα χαρακτηριστικά της νομίζω ότι καθιστούν ιδεώδη υποψήφιο. Πέραν αυτών, η θετική ψήφος προς την κυρία Μπετίνα Ιάκοψεν ε, λαμβάνει υπόψη και το γεγονός ότι θα είναι η πέμπτη, ε, το πέμπτο μόνο μέλος γυναίκα του ελεγκτικού συνεδρίου. Πρέπει λοιπόν να σημειώσουμε ότι χρειάζεται περισσότερη εξισορρόπηση της εκπροσώπησης των φίλων στο ελεγκτικό συνεδρίο κυρία Ιάκοψεν έχει στρατευτεί και εκδηλώσει την αφοσίωσή της στην ε, ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Ελεγκτικού Συνεδρίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κυρίως Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού με βάση και την ε, διαδικασία που προβλέπεται από τα νομοθετήματα τα σχετικά με τη διαχείριση του προϋπολογισμού και τον ελεγχό της εκτέλεσής του. Πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε μια πιο πλήρη επισκόπηση της σταδιοδρομίας των ελεγκτών, των μελών δηλαδή του Ελεκτικού συνεδρίου στο μέλλον, ώστε να μπορούμε να κρίνουμε πιο ουσιαστικά. Μας έχει πει η κυρία Μπετίν Άντερσεν ότι θέλει πιο αποτελεσματική διαχείριση και του, της διαδικασίας ελέγχου και εγώ ίδιος ως πρώην επικεφαλής του ελεγκτικού συνεδρίου της Δανίας και γνωρίζοντας τη σταδιοδρομία της κυρίας Γιάκοψεν θα ήθελα να εκφράσω την πλήρη υποστήριξή μου και να πω στο σώμα ότι προτείνω να υποστηριχθεί η υποψηφιότητά της ως νέου μέλους από τη Δανία στο ελεγκτικό συνέδριο. Ευχαριστώ πολύ. Πρόκειται για μία και μόνο ψηφοφορία, μυστική για την υποψηφιότητα αυτή. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται η υποψηφιότητα. Ο διορισμός καλύτερα. Έκθεση Μαστάλκα. Άσκηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση των δικαιωμάτων από το Διεθνές Εμπόριο. Παρακαλώ, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση Μαστάλκα και πάλι άμυνα κατά τη ζημιογόνου τιμολόγηση των πλοίων. Μία και μοναδική ψηφοφορία ονομαστική. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση Φεραίρα. Αλληλευτικές δυνατότητες ενωσιακά ύδατα σε αλληλευτικά σκάφη που φέρνουν σημαία τη βολιβηριανή δημοκρατία τη Βενεζουέλα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη στα νικά των ακτών τη Γαλλική Γουινέα. Μου θέλετε το λόγο, κύριε συνάδελφε, όχι. Παρακαλώ. Μάλιστα, εδώ και αρκετά χρόνια τα σκάφη της Βενεζουέλα αλλιεύουν στα ύδατα της Γαλλικής Γουινέας, ε, ε συγγνώμη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να ε, το σταματήσουμε για να αναπτυχθεί η απασχόληση στην Γαλλική Γοιάννα. Θα πρέπει λοιπόν να προστατευτούν. Δεν υπάρχει λόγος για θεσμική, ε, θεσμικό τσακωμό ή σύγκρουση. Ε, έχει επιληθεί το θέμα, έχει ξεπεραστεί αυτή τη στιγμή από το Συμβούλιο και αυτό που προτείνουμε είναι όσο γίνεται πιο σύντομα να μπορέσουμε να εγκρίνουμε αυτή τη σύσταση. Είναι σημαντικό να πούμε ότι η Βολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας θα πρέπει να σεβαστεί όλες τις συμφωνίες ε, που έχει αναλάβει, όλα μάλλον τις διατάξεις που έχει αναλάβει με αυτήν την ε, συμφωνία και την αναφορά των, των αλλιευμάτων, πράγματα ε, τα οποία ισχύουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό το λόγο πρέπει να εγκριθεί αυτή η σύσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και ψηφίζουμε μοναδική ψηφοφορία ονομαστικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Έκθεση Κάρτια Σαββάλου Ρουμπιάλ, σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού υπαριθμών 3 στο Γενικό Προπολογισμό του 2015, γραφή του Πλεονάσματο Οικονομικού του 2014, ονομαστική ψηφοφορία μοναδική, αρχή ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Και συνεχίζω με την κυρία Καρδιά Ζαβάλ Βιάλα. διορθωτικός προπολογισμό για την κινητοποίηση του Ταμείου Ελέγγυη τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Ιταλία. Μοναδική ψηφοφορία. Ονομαστική. Άρχεται. Πέρα. Εγκρίνεται. Έκθεση Μπουρεσάν. Συνειδητοποίηση Ταμείου Ελεγγύη Ευρωπαϊκή Ένωση πλημμύρε στη Ρουμανία, την Βουλγαρία και την Ιταλία. Μοναδική ψηφοφορία ονομαστικά. Αρχίζει. Πέρας. Έκθεση ΚΟΧ. Παροχή ολοκληρωμένη πολυτροπική έκδοση εισιτηρίων στην Ευρώπη. Μοναδική και ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Μου ζητήθηκε δυνάμει το άρθρο 197 του κανονισμού από τη διάσκεψη των Προέδρων να ε, ψηφίσουμε την παράταση της θητεία τη Ειδικής Επιτροπή για τις Προγραμματικές Αποφάσεις τύπου tax ruling και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος έως τις 30 Νοεμβρίου του 2015, αν δεν έχουν, ε, αν δεν έχουν εκφράσουν Εγκρίνεται αυτή η παράταση, δεν βλέπω αντιρρήσει. Εγκρίνεται λοιπόν και έτσι περνώ στην έκθεση Καρδιά Βάλου Ρουβιάλ πάλι. Σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων έτσι ονομαστικά μοναδική ψηφοφορία, αρχική ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε την κυρία Καρδία Ζαβάλ Ρουβιάλ, σχέδιο ορθωτικού προπολισμού, αντιμετώπιση των μεταναστευτικών πιέσεων. Μοναδική και ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση Νίκολσον επανεξέταση της εφαρμογής της μέτρων για το γαλακτοκομικό τομέα. Ποιο είστε στο λόγο, Αλήθεια, Παρακαλώ, κυρία μου. Έχουμε ένα θέμα εδώ. Θα ήθελα να δοθεί κάποια διευκρίνηση, γιατί έχουμε μια τροπολογία που είναι σημαντική και δεν είμαι σίγουρη τι ακριβώς σημαίνει. Έχουμε την 22. Θα ήθελα να μου πείτε αν πράγματι η αυτό σημαίνει πως είμαστε υπέρ ή κατά των ποσοστώσεων στο γάλα. Θα ήθελα να μου το εξηγήσετε γιατί από αυτό εξαρτάται το πώς θα ψηφίσουμε. que 6, Παράγραφος 6, αρχικό κείμενο, ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 9 αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές θα πρέπει να το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά, παρακαλώ πολύ, για την παράγραφο 9 θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, ξεκινά. Λίγη. Εγκρίνεται. Παράγραφος 10. Αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15. Αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 22. Αρχικό κείμενο είναι ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη. Απορρίπτεται. 24 αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Θα πρέπει να επαληθεύσουμε λοιπόν ηλεκτρονικά για την 24. Αρχίζει. Λίγη απορρίπτεται. 26 αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές και πάλι δεν το καταλαβαίνω επαλήθευση ηλεκτρονική για την παράγραφο 26 αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη. Εγκρίνεται. 36 αρχικό κείμενο υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται 47 αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές δεν εγκρίνεται. Νομίζω θα επαληθεύσουμε γιατί 54 ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγοι. Εγκρίνεται. 42 υπέρ. 62 με συγχωρείτε υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 66 ονομαστικά αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη. Εγκρίνεται. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 69. Ονομαστικά αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη. Εγκρίνεται. 70 σε δύο τμήματα για το πρώτο ποιος είναι υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά απορρίπτεται 72 στο κείμενο μας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται στο ε, εκτιμώντας στην σκέψη ε, J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα, ολόκληρο το ψήφισμα, ηλεκτρονικά, ονομαστική ψηφοφορία, αρχίζει ψηφοφορία. Λίγη. Εγκρίνεται. Μπορούμε τώρα να περάσουμε στην έκθεση Ζαραντίλα ο εξωτερικός αντίκτυπος εμπορικής και επενδυτικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τρίτες χώρες. Έχουμε ε, μία συνάδελφο που θέλει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας πω το εξής. Εγώ δεν ξέρω αν δεν κατάλαβα εγώ ή, ή αν έπρεπε να έχουμε κάνει ένα λεπτό σιωπής για τα θύματα της ε, τρομοκρατικής επίθεσης όπως ζήτησαν δύο μέλη του Κοινοβουλίου. Νομίζω χρόνο έχουμε. Ένα λεπτό ζυγής μπορούμε να τηρήσουμε. Μπορούμε να διαθέσουμε ένα λεπτό του χρόνου μας για το ζήτημα αυτό. Δεν θα θυσιάσουμε χρόνο. Δεν ήταν εκεί το πρόβλημα ότι λείπει ο χρόνος. Εάν θέλετε λοιπόν τώρα ένα λεπτό σιγής για τα θύματα αυτά. Merci. Reprenons donc le Ωραία λοιπόν. Προχωράμε στην έκθεση Ζαραντήλ και έχουμε μια πρόταση εδώ αντικατάστασης ε, που θα ψηφίσουμε. Η Γκουέ έχει υποβάλει αυτή την πρόταση. Υπέρ της πρότασης Γκουέ λοιπόν εδώ ποιος είναι. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Περνάμε λοιπόν στην παράγραφο 9. Υπέρ. Α, είναι σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω απορρίπτεται, αλλά θα ήθελα να επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά για το δεύτερο τμήμα της 9 παραγράφου. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη. Εγκρίνεται. Ωραία, λοιπόν, ολόκληρο το ψήφισμα. Ονομαστικά ε, αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη. Εγκρίνεται. Περνάμε λοιπόν στην έκθεση μέλο για τον τομέα των οροκυπευτικών από τη μεταρρύθμιση του 2007 έως σήμερα. Παράγραφος 18 του κειμένου μας. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 59 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 60 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται ολόκληρο λοιπόν ε, ονομαστικά αρχίζει η ψηφοφορία για ολόκληρο το κείμενο λίγη εγκρίνεται ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι θα περάσουμε τώρα στις επεξηγήσεις ψήφου